you, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων ζήτησε να λάβει περαιτέρω πληροφορίες από τον υποψήφιο Επίτροπο κύριο Χιλ ώστε να περατωθεί η αξιολόγησή της του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίτροπος έχει δώσει απαντήσεις σε μια σειρά πρόσθετων γραπτών ερωτήσεων και στη σημερινή συνεδρίαση θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων, μια πρόσθετη ακρόαση για τα θέματα αυτά που ήταν το αντικείμενο των ερωτήσεων ώστε να υπάρξουν διευκρινήσεις που δόθηκαν γραπτά. Έχουμε μονάχα μια μισή ώρα για την ακρόαση αυτή, την πρόσθετη ακρόαση. Θα ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν την αρχή των ε, χρονοθυρίδων τριών λεπτών και υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι ο στόχος σημερινής ακρόασης είναι να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα τα οποία ηγέρθησαν στις πρόσθετες ερωτήσεις μας. Είναι λοιπόν για τις πρόσθετες αιτήσει διευκρίνησης, όχι για γενικά θέματα. Δίνω λοιπόν <clears throat> καταρχήν το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο κύριο Χιλ για την εισαγωγική του παρέμβαση 10 λεπτών και μετά θα έχουμε 24 ε, ερωτήματα, 3 λεπτών το καθένα, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο για την απάντηση και στη συνέχεια ο υποψήφιος επίτροπος έχει 3 λεπτά για μια καταληκτική παρέμβαση. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χιλ για την ε, εναρκτική του, εναρκτήρια του παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ. Όταν σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι προσέβλεπα να σας στην ε, επόμενη συνάντησή μας, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Στα αγγλικά πρέπει να προσέχει κανείς τι εύχεται γιατί μπορεί να του έρθει στο κεφάλι. Εδώ είμαι πάντως ενώπιόν σας. Χαίρομαι που έχω επιστρέψει ενώπιόν σας. Και είναι κατά κάποιο τρόπο μια προκαταβολή αυτών που ελπίζω να γίνουν στο μέλλον, δηλαδή μιας καρποφόρας και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ μας. Νομίζω ότι έχετε δει τις απαντήσεις μου, τις λεπτομερείς απαντήσεις στα 23 πρόσθετα ερωτήματα που θέσατε. Καταρχήν όμως θα ήθελα να κάνω, αν μπορώ, ένα βήμα πίσω και να σας ζητήσω να φανταστείτε ότι είναι το 2019. Βρισκόμαστε ενώπιον των επομένων ευρωεκλογών και φτάνουμε στο τέλος της θητείας της Επιτροπής Juncker. Η προς το τέλος της ε, θητείας της πρώτης Επιτροπής γιονκερ; Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που μπορούμε να δώσουμε στους ψηφοφόρους μας. Τι πετύχαμε με τη συνεργασία μας για τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Η συνολική λοιπόν εικόνα για το 2019 θα είναι η Ευρώπη γύρισε στην ανάπτυξη. Μειώνεται η ανεργία, ιδίω η ανεργία των νέων. Οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που πέρασαν πολλές χώρες, ιδίως στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ευρώπης. Οι κρίσεις αυτές έχουν περατωθεί, έχουν τελειώσει. Γυρίζουν οι χώρες αυτές σε οικονομική υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρότερη και πιο συνεκτική και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και πολιτικές ανησυχίες των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά παραμένει μια οικογένεια 28 κρατών μελών μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε εκ νέου επιτύχει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μια ισχυρή τραπεζική ένωση που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια ισχυρότερη και καλύτερα διαχειριζόμενη ζώνη του ευρώ και έχουν δώσει μεγαλύτερη ακτινοβολία στο ευρώ σαν παγκόσμιο νόμισμα. Με την υποστήριξη της Κομισιόν, όλο και περισσότερα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην Τραπεζική Ένωση. Η εμπιστοσύνη χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτών που είναι μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην ε, ε, Τραπεζική Ένωση, μάλλον και αυτών που δεν είναι μέσα, επί τη βάση ενό κοινού ε, βιβλίου κανόνων για τα τραπεζικά θέματα. Καμιά τράπεζα δεν είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να επιτραπεί η αστοχία της. Έχουμε εξασφαλίσει την πολυμορφία του τραπεζικού συστήματος. Έχουμε και πάλι τράπεζες με ισχυρότερου ισολογισμού και που δανείζουν στην υπόλοιπη οικονομία γιατί έχουμε εξασφαλίσει τι σωστέ διαρθρωτικές αλλαγές. Οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στις τράπεζες και στην ασφάλεια των καταθέσεών τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζεται ως ένας ε, επόπτης παγκόσμιας εμβέλειας. Οι δοκιμασίες αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής την χάνουν εμπιστοσύνη και δίνουν μια σωστή ανάλυση τη υγεία των τραπεζών. Οι καταναλωτέ χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη επιλογή ασφαλέστερων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε χαμηλότερο κόστο όπω συντάξει και ασφαλίσει. 60 χρόνια μετά από την έγκριση της συνθήκης της Ρώμης, επιτέλους βλέπουμε την ανάδυση μιας ενιαίας αγοράς κεφαλουχικών προϊόντων. Την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Έχουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που προστατεύει τους καταναλωτές και τους επενδυτές και δίνει εμπιστοσύνη και σωστό πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη, καλά διαχειριζόμενη, διάφανη και ρευστή αγορά κεφαλαίων σε όλα τα κράτη-μέλη Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά η Ευρώπη χαίρεται και είναι υπερήφανη για το σύστημα χρηματοπιστωτικών τη υπηρεσιών που εμποδίζει ανεύθυνη ανάληψη κινδύνου και βραχή ε, βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση, όπω έγινε στο παρελθόν, αλλά επιτρέψει στι εταιρείε να, ε, να καινοτομούν και να επενδύουν με σόφρονα τρόπο μακροπρόθεσμα. Επίση, χαιρόμαστε για το ρόλο μα στη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενό στεναρού συνόλου διεθνών κανόνων για τι χρηματαγορέ, που αναγνωρίζονται από όλους και ιδίως στις ταχαίως αναδυόμενες οικονομίες. Πάνω απ' όλα, το 2019 θα είμαστε υπερήφανοι για το ρόλο μας στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επί τη βάση της αξίας τους και όχι επί τη βάση της χώρας στην οποία λειτουργούν. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές που δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, αντιμετωπίζουν τις μεγάλες εταιρείες και με το να διαμφισβητούν το status quo κάνουν την οικονομία μας και την κοινωνία μας πιο ασφαλή. Και είναι οι πολίτες οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα κερδίσουν περισσότερο από την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξαναγυρίζω όμως το 2014. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι θα, δεν θα υπάρξουν δυσκολίες στον δρόμο μπροστά μας. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν ε, απόψεις για τις οποίες είναι απόλυτα πεπισμένοι και επιχειρηματολογούν υπέρ αυτών. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, γιατί πολλά από τα δομικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για το μέλλον αυτό υπάρχουν ήδη. Αν συνεργαστούμε και παραμείνουμε πιστοί στην πορεία μας, πιστεύω μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική, σταθερή και παγκόσμια ανταγωνιστική ε, ε, περιοχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ένα κλάδο ο οποίος θα μπορεί να χρηματοδοτεί τη μακροχρόνια ανάπτυξη και δίνει περισσότερα ωφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή αυτή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για τη μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε μια μεγάλη συνεισφορά στην Ευρωζώνη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Πράγματι όλα αυτά θα απαιτήσουν σημαντική κοινή εργασία. Γνωρίζω όμως ότι η Επιτροπή σας είναι συνηθισμένη σε αυτή τη συνεργασία. Θέλω να, να συνεχίσω το έργο του Μισελ Μπαρνιέ, να δημιουργήσω ε, εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και φυσικά και με τα κράτη-μέλη. Εάν με εγκρίνετε στο αξίωμα αυτό από την 1η Νοεμβρίου, έχω να σας δώσω μια απλή υπόσχεση. Θα είμαι ένας Ευρωπαίος Επίτροπος και για όλες τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεργαστώ μαζί σας όσο μπορώ πιο σκληρά και όπως ξέρω να εργάζομαι για να μπορέσω να κάνω αυτό το όραμα πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Υποψηφιέ Επίτροπε. Υπενθυμίζω τους, στους συναδέλφους ότι έχει απαντήσει γραπτό ο υποψήφιος επίτροπος ε, σε 23 ερωτήσεις και τώρα να αρχίσουμε και ο πρώτος ομιλητής μας θα είναι ο Παύλος Αμπαμπίντεκαν. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επίτροπο. Έχω δύο ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά το στόχο σας να εξασφαλίσετε πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Φυσικά συμμερίζομαι πλήρως αυτό το στόχο και πιστεύω ότι ακριβώς για να το πετύχουμε θα πρέπει να υλοποιήσουμε την Ένωση των Αγορών. Μπορείτε να μας συγκεκριμενοποιήσετε τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την Ένωση των Αγορών. Δεύτερον, για το TTIP, τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συμπερίληψη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στι διαπραγματεύσει. Βέβαια δεν εμπίπτει αυτό στι δικέ αρμοδιότητε, αλλά οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε ανήκουν στον τομέα διαπραγματεύσεων του TTIP. Σκοπεύετε να εξασφαλίσετε συμπερίληψη στι διαπραγματεύσει των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Δύσκολο είναι να απαντήσω ενδελεχώ και στι δύο ερωτήσει για το TTIP. Είναι σημαντικό το είδος της συνεργασίας που θα έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να περιχαρακώνεται βέβαια από την TTIP, αλλά θέλουμε ένα συγκεκριμένο και στιβαρό πλαίσιο. Τώρα για την Ένωση των Κεφαλαίων νομίζω ότι είναι από τις πιο συναρπαστικές ευκαιρίες που έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι η συνολική μας στόχη είναι να έχουν οι επενδυτές να τύχουν τι δέωσες προστασία και να έχουν εμπιστοσύνη στι επενδύσει, να προσελκύσουμε επενδυτέ και επενδύσει από όλο τον κόσμο και φυσικά να θαρρύνουμε την ελεύθερη ροή κεφαλαίων. Και για να το επιτύχουμε θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά μέσα, να τονώσουμε την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλο μακροπρόθεσμο και μεγάλη πίβολο σχελίο. Θέλουμε να ευαθύνουμε τι εργασίε για το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, σημαντικό αυτό και θέμα του δικαίου αφαιρεγκαιότητα και του εταιρικού δικαίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θέλουμε ενίσχυση του, του ε, εποπτικού πλαισίου και εφαρμογή του. Τώρα, έχουμε τρεις τομείς ε, που χρήζουν άμεσης δράσης. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε το συντομότερο δυνατό την πρόταση για το ΕΛΤΙΦ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων, ώστε να ε, μπορέσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το θέμα της οδηγίας προσπέκτους για τα ενημερωτικά δελτία και αυτό θα επηρεάσει θετικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης με τη MIFID 2 και θα έχουμε νέες ευκαιρίες ε, για ανάπτυξη και πραγματοποίηση συγκεκριμένων βημάτων. Όπως είπα και στην προηγούμενη ακρόαση και πριν από λίγο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ενδελεχή ανάλυση και διάγνωση των προβλημάτων. Και εντόπισα στην ανάλυση κάποιους φραγμούς και εμπόδια, να αναλύσουμε τα προβλήματα, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να υλοποιήσουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Η κυρία Ελίζα Φερέιρα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που ξανά ήρθατε. Στις γραπτές απαντήσεις, κύριε Υποψήφιο Επιτροπέ, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι ένα ενιαίο καθεστώς εγγύης καταθέσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, επιθυμητό. Αυτό αναφέρει η Επιτροπή στις δηλώσεις της. Είπατε όμως ότι φαίνεται ότι δεν έχουν οριμάσει πολιτικές συνθήκες για μια τέτοια αλλαγή. Βέβαια, θα εξετάσετε κάποιε αναλλακτικέ λύσεις μετά τον Ιούλιο του 2019 για το ισχυρό σύστημα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως περιχαρακώνεται από τι συνθήκες, ε, δεν είναι να περιμένει τι προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά να αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία εξυπηρετώντα του πολίτε και το κοινό συμφέρον. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είστε έτοιμος να διαδραματίσετε το θεσμικό σας ρόλο και να υλοποιήσετε τις υποσχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλοντας σχετική πρόταση για ένα ενιαίο κοινό σύστημα ε, εγγύησης των καταθέσεων πριν το 2019. Ναι, γνωρίζω πόσο προσφυλέ σα είναι το θέμα αυτό. Τώρα, καταρχήν πριν από λίγους μόνο μήνες αποφάσισαν ε, οι συνομοθέτες να μην υιοθετήσουν ένα ενιαίο καθεστώς εγγύηση των καταθέσεων. Έχουμε μια πολύ πρόσφατη απόφαση για το θέμα αυτό. Αυτό είναι το σημείο εφετηρίας. Τώρα, ως προς την αρχή. Όπως φαίνεται και από την απάντησή μου, ένα ενιαίο καθεστώς ε, εγγύηση των καταθέσεων είναι ε, μακροπρόθεσμα ένας, πιο, ένας αυτονόητος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Αν είχαμε ξεκινήσει εκ του μηδενός, ε, που θα ήταν λογικό, δεν θα, θα το κάναμε. Αλλά δεν ξεκινήσαμε εκ του μηδενός. Έχουμε ένα εφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο σεβόμαστε. Και ο προκάτοχός μου προτίμησε την εναρμόνιση πρώτα για τις εγγύησεις καταθέσεων. Και νομίζω ότι δεδομένου των συνθηκών και των πολιτικών ε, καταστάσεων είναι μια λογική επιλογή. Τώρα, με ρωτήσατε αν θα πρέπει να περιμένω το 2019 που είναι η ημερομηνία που προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση. Από τη στιγμή που έχουμε λειτουργικές, ε, ε, λειτουργική καθεστώτα εγγύης καταθέσεων μαζί με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και το ενιαίο το μηχανισμό εξυγίασης θα έχουμε πιο πρόσφορες συνθήκες και τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν και σίγουρα οι κανόνες θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί όπως ε, επισημάνατε κι εσείς. Αφού λοιπόν πληρωθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα δούμε πώς λειτουργεί η οδηγία αυτή για τις εγγύησεις καταθέσεων και μαζί με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα εξετάσουμε το θέμα και ίσως υποβάλουμε κάποιες προτάσεις πριν τον Ιούλιο του 2019. Πάντως, δεδομένων των σημερινών περιστάσεων και συνθήκων, κρατούμε το θέμα ανοιχτό, θα το επανεξετάσουμε και θα το συζητήσουμε και μαζί. Και ίσως νωρίτερα και από τον Ιούλιο του 2019. Ευχαριστώ. Κέιτ Σουίνμπορν από την ομάδα συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε και πάλι κύριε Χιλ. Η ομάδα μου δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να επανέλθω. Νομίζω ότι και την πρώτη φορά τα πήγατε εξαιρετικά. Οι ερωτήσεις μου θέλουν να σας βοηθήσουν να τηρήσετε το χρόνο. Ξέρω ότι σε δύο λεπτά είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς πλήρη απάντηση. Παρακαλώ, μήπως μπορείτε να πείτε περισσότερο για το πώς θα βοηθήσετε τις μικρομεσαίες να αναπτυχθούν. Πολλοί ασχοληθήκαν πολύ με τη MIFID και την αναθεώρηση της MIFID οδηγίας. Πέστε μας, πώς θα, η αγορά για την ανάπτυξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων πώς θα είναι προσβάσιμη και για τους καταναλωτές και για τους επενδυτές. Ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίδετε. Όπως είπα και προηγουμένως, χαίρομαι πολύ που ήρθα και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Τώρα, τι συγκεκριμένα μπορούμε να κάνουμε για την ε, αντίληψη αυτή για μια ε, αγορά ανάπτυξη των μικρομεσαίων και την αντίληψη αυτή ανάπτυξη των μικρομεσαίων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε φυσικά τις μικρομεσαίες για μια σειρά από λόγους. Θα είναι προτεραιότητα κλειδί, απόλυτη προτεραιότητα κλειδί για όλους τους τομείς ανασχόλησής μου. Τώρα από πού θα υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι από τράπεζες ή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης αλλά με βάση την Ένωση Κεφαλαιαγορών πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση. Όπως ξέρετε καλύτερα από πολλούς, επειδή ξέρω ότι ασχοληθήκατε πολύ με τη MIFID 2, εισάγουμε την έννοια αυτής της αγοράς ανάπτυξης των μικρομεσαίων, που είναι μια δυνατότητα όπου μπορούν να γίνουν συναλλαγές, ε, όπου η μισή από αυτούς που θα εκδίδουν τίτλους είναι μικρομεσαίες, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς χωρίς βαριές ρυθμίσεις για να ενθαρρύνουμε τις ε, ροές επενδύσεων. Οι λεπτομέρειες φυσικά θα συμπεριληφθούν σε μία κατεξοδότηση πράξη. Για τις λεπτομέρειες δεν μπορώ παρά να πω με χαρά θα συνεργαστώ και με εσά και με άλλους που γνωρίζετε τον τομέα για να δούμε πώς μπορούμε όντως να διαμορφώσουμε το κείμενο αυτό, αλλά πιστεύω ότι αν επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των τμήματων του κειμένου, θα βοηθήσουμε πολύ την οικονομία, όπως είπα και προηγουμένως, οι μικρομεσαίες που κάνουν αυτό το πρώτο βήμα, να προσπαθήσουν να ε, εκδώσουν τίτλους για να βρουν χρηματοδότηση, δεν μπορούν να έχουν ε, πολλές υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ε, για παράδειγμα, τι είδος λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλουν, ποιος θα τους ελέγξει. Το βασικό είναι αυτή η ιδέα για μια ε, αγορά ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκουλάρα από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Λόρδε Χίλ που επανήλθατε ενώπιόν μας. Ευχαριστώ για τις αναλυτικές απαντήσεις σας. Ε, πραγματικά σοβαρά αντιμετωπίσατε την ακρόασή σας και το εκτιμούμε. Μία ερώτηση, τώρα που έχουμε πιο αναλυτικές απαντήσεις. Μία ερώτηση που είναι ανάμεσα στις απαντήσεις σας 11 και 12. Εγώ αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Με ακούτε, με ακούτε. Ξαναρχίζω, ξαναρχίζω. Ξαναρχίζω, ξαναρχίζω. Εντάξει, εντάξει, με ακούσατε, με καταλάβατε. Ωραία. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν, η ισχύ της Ευρώπης στον κόσμο είναι για μένα μεγάλη ανησυχία μεταξύ των απαντήσεων σας 11 και 12 ε, είναι η αντιμετώπιση λίγο ελαφρώς διαφορετική να ε, εξετάσω αν συμφωνούμε για την ε, απάντηση στο 12. Φυσικά πρέπει να υπάρξει συναρμόνιση των κανόνων μας με άλλα τμήματα του κόσμου, τους Αμερικανούς, τους Κινέζους, τα... εντός του G20. Και αυτό κράτησα εγώ από την απάντησή σας και θέλω να είμαι σίγουρη ότι όντως ισχύει, είστε όντως δεσμεύεστε να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα της Ένωσης, γιατί δεν είμαστε πάντα στο ίδιο μήκος κύματος. Για... Το να λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε καταστάσεις τραπεζικών τομέων πολύ διαφορετικών μου φαίνεται λίγο επικίνδυνο. Να πούμε λοιπόν ότι φυσικά θα συνεργαστούμε με τους άλλους και θα το συζητάμε συχνά, αλλά συμφωνείτε απόλυτα ότι πρέπει να υπερασπιστείτε το γεγονός ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες και το κύριο δεν είναι να αρμονίσουμε τους κανόνες, αλλά να καταλήξουμε μαζί με τους άλλους σε δίκαιες λύσεις. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, δεν είχα διαλέξει το σωστό κανάλι. Ε, αλλά έτσι τα γυμνασιακά γαλλικά μου έδειξαν πόσα αξίζουν. Βεβαίως, βεβαίως, ε, οι ιδιαιτερότητες μας είναι σαφείς και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι πάντα πρέπει να στοχεύουμε σε πλήρη ταυτότητα κανόνων. Βεβαίως, στόχος μας πρέπει να είναι να υπάρχει ισοτιμία, ισοδυναμία των κανόνων. Επίσης, να καταλάβουμε τη θέση μας. Γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε σε όλους ακριβώς τους ίδιους κανόνες, γιατί αυτό μπορεί να επιβραδύνει την ε, επιτυχία των προσπαθειών μας. Η ισοδυναμία είναι η σωστή προσέγγιση. Πρέπει στόχος μας να είναι τα αποτελέσματα και να υπάρχει προληπτική αντιμετώπιση. Δεν θεωρούμε ότι οι άλλες δικαιοδοσίες πρέπει να έχουν ακριβώς ε, τους ίδιους κανόνες, γιατί και το νομικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές του κόσμου αλλά οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε πολύ αυστηρή τεχνική αποτίμηση των κανόνων των τρίτων χωρών. Μόνο αν μπορούμε να σεβαστούμε την τρίτη χώρα μπορούμε να αφαιθούμε στην εφαρμογή των δικών της κανόνων και της δικής της εποπτείας. Αυτός πιστεύω είναι ο καλύτερος τρόπος να υπάρξει πραγματική ουσιώδης και αποτελεσματική εποπτεία. Πρέπει να είναι ισοδύναμη και φυσικά δεν είναι μονόδρομος τίποτα. Οι άλλες ε, περιοχές πρέπει να έχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να αναγνωρίζουν την ε, ισχύ των δικών μας κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω θα επιχειρήσω να ε, προωθήσω το θέμα αυτό στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι συμφωνείτε πως αυτή είναι συγκεκριμένη αντιμετώπιση που στοχεύει στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Κύριε ναι. Χίλ, ε, στις ερωτήσεις που σας ε, στείλαμε, εσείς πάλι αρνηθήκατε να απαντήσετε ε, στο θέμα των ε, οργανισμών υπέρ των οποίων είχατε ασκήσει λειτουργία ως λομπίστας στο παρελθόν. Είπατε ότι έχει περάσει η εποχή των περιστρεφωμένων θυρών. Αλλά εσείς έχετε περάσει τόσες φορές αυτές τις περιστρεφόμενες θύρες που ίσως έχετε ξεχάσει τι έχετε κάνει. Μπορεί το Κοινοβούλιο να πιστεύει ότι δεν θα επιστρέψετε σε αυτό το παρελθόν όταν ασκείτε το λειτουργήμα του Επιτρόπου. Και δεύτερον, τα θέματα διαφάνειας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένας επίτροπος με τη δική σας ευθύνη θα πρέπει να εξασφαλίσει κυρίως την, την διαφάνεια έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς περιμένετε λοιπόν ότι αυτό το Κοινοβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα επίτροπο ο οποίος αρνείται με τοπικά να απαντήσει στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου για το έργο του λομπίστα στο παρελθόν. Uh, first of all... Πρώτα απ' όλα, για τη διαφάνεια. Και πώς πρέπει να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο και με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζω ότι κατάφερα στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε συνολογικά στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων να τονίσω πόσο σοβαρά παίρνω αυτό το θέμα της διαφάνειας και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνει κανείς αυτό πραγματικότητα σε σχέση με τη δημοσιότητα των συναντήσεων και των πορισμάτων τους, σε σχέση με το να εξασφαλίσω ότι φορείς οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε ομίλους μεγάλων επιχειρήσεων δεν συνδέονται με αυτούς είναι σε θέση να διαμφισβητήσουν την κρατούσα άποψη το να υπάρχει ένα υποχρεωτικό μητρό για το οποίο ανέφερε ο κύριος Γιούνκερ για τα λόμπι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξασφαλίσουμε λοιπόν την διαφάνεια. Για μένα προσωπικά, γιατί αυτό ήταν και το πρώτο σας ερώτημα, Ίσως εδώ πρέπει να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ως λομπίστα, όταν ήμουνα στη Βουλή των Λόρδων, έκανα πιο σφιχτούς και πιο αυστηρούς τους κανόνες για τα λόμπι. Και ο λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσα να σας δώσω απάντηση στα ερωτήματά σας, και αυτό δεν είναι έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο, είναι απλώς δήλωση μιας πραγματικής κατάστασης. Οι εταιρείε αυτές που εργάστηκα εκεί πριν από 25 χρόνια έχουν αλλάξει χέρι, έχουν αλλάξει διοίκηση. Δεν έχω τη δυνατότητα να ξέρω τι πληροφορίε υπάρχουν ακόμα για τα θέματα αυτά. Για αυτό το θέμα του για ποιους εργάστηκα στο παρελθόν, που είναι ένα λογικό ερώτημα, πρέπει να σας πω ότι πριν από 4,5-5 χρόνια έπαυσα να εργάζομαι με οποιαδήποτε εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είχα καμία σχέση με καμία από τι εταιρείε στι οποίε εργάστηκα επαγγελματικά ή συνδέθηκα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν είχα καμία τέτοια σχέση μαζί του, δεν άσκησα καμία δραστηριότητα λόμπι στα ευρωπαϊκά όργανα σε αυτό το διάστημα. Επομένω το ερώτημα πρέπει να είναι αν έχω κάποιο κίνητρο ή κάποια θέληση να παίξω το ρόλο αυτό του λομπίστα, εγώ παίρνω πολύ στα σοβαρά την νομική μου ευθύνη, παίρνω πολύ σοβαρά την ε, δέσμευση που παίρνω ως Επίτροπος προσωπικά και θεσμικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ακολουθεί ο Σβέν Γκίγκολτ από τους Πράσινους. Λόρδε Χίλ, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή στο παραμύθι κατά κάποιο τρόπο που μας αναφέρατε για το 2019. Και είναι πολύ ωραία η φωνή σας και ο τρόπος με τον οποίο να φυγηθήκατε αυτό το παραμύθι. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται και μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον για να ακούσει ένα παιδάκι. Αλλά πέραν αυτού, από τη δική μου οπτική γωνία νομίζω ότι δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνη στο οποίο τίθεται. Το ερώτημα είναι αν εσεί με το παρελθόν σα, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η υποψηφιότητά σας, Ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί θέματα εμπιστοσύνης. Ένα μονάχα παράδειγμα. Για τις εταιρείε που εργαστήκατε δεν μας είπατε ούτε μία τέτοια εταιρεία. Αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Δεν μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα εταιρεών για τις οποίες ασκήσατε δραστηριότητα λομπίστα. Αυτό θα μας έδινε την εντύπωση ότι θέλετε να σπάσετε τη σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίσατε τη δουλειά στο παρελθόν και ότι έχετε μια νέα προσέγγιση τώρα. Λυπάμαι, λέει ο Λόρδος Χιλ, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε το θέμα της ε, εμπιστοσύνη. Έχουμε συζητήσει και προσωπικά για το θέμα αυτό και σας εξήγησα τα πράγματα όσο μπορώ πιο σαφώς. Στην απάντησή μου αναφέρθηκα στις εταιρείε στην Quilliam, όπου ε, είχα εργαστεί στο παρελθόν. Όλα αυτά είναι, είναι δημόσια γνωστά, ότι εργάστηκα εκεί μέχρι να φύγω. Όλα αυτά μπορεί να τα δει οποιοδήποτε. Και για αυτούς που ενδιαφέρονται λοιπόν, μπορώ να είμαι απόλυτα σαφής, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, η πλευρά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αυτής της επιχείρησης δεν ήταν ένας τομέας με τον οποίο εγώ είχα εμπλακεί ιδιαίτερα. Το τμήμα αυτό που έχει να κάνει με τις δημόσιες σχέσεις, το τμήμα που θα ονομάζατε εσείς lobbying, ήταν μονάχα ένα μικρό κομμάτι της, ε, εταιρείας. Η εντύπωση λοιπόν η οποία δημιουργήθηκε ότι εγώ βρισκόμουν στην τσέπη μέσα σε εισαγωγικά πολλών μεγάλων εταιριών στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ότι περνούσα περιστρεφόμενες θύρες, αυτό δεν είναι σωστό. Έφυγα σχεδόν πέντε χρόνια πριν για να μπορέσω να μπω στο δημόσιο τομέα και αυτή η περίοδος της ζωής μου, για την οποία εγώ είμαι υπερήφανος, γιατί νομίζω ότι δημιούργησα μια επιτυχή επιχείρηση, ήμουν καλός εργοδότης και λειτουργήσα αυτή η επιχείρηση πολύ καλά. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν, δεν έχω καμία πρόθεση, καμία επιθυμία να επανέλθω. Έχω ακολουθήσει το δρόμο του να είμαι ε, δημόσιος αξιωματούχος, υπουργός, να μπορέσω να κάνω πράγματα στον τομέα της παιδείας και τώρα ως επίτροπος στην Ευρώπη. Για να είμαι λοιπόν ειλικρινής, όλα αυτά δεν έχουν πραγματική υπόσταση. Δεν θα κάνω απολύτω τίποτα το οποίο θα κυλιδώσει το κύρος και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα δημιουργήσω τέτοια προβλήματα. Είμαι έτοιμος να εργαστώ με απόλυτη ακαιρεότητα για το λειτουργήμά μου. Ευχαριστώ για την ομάδα EFDD Steven Wolf στην εισαγωγική ομιλία σας είπατε ότι το μέλλον θα είναι λαμπρό για την Ευρώπη. Το περιγράψατε. Είστε υποψήφιος επίτροπος και λόρδος. Τώρα έχετε γίνει και η πυθία της Ένωσης. Είπατε ότι οι οικονομίες της Ευρώπης θα τα πάνε καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα είπατε τι θα σας πει η Βασίλισσα για τον όρκο σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ομιλία σας είπατε ότι ότι η Ένωση θα παραμείνει με 28 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί αν γίνει δημοψήφισμα, θεωρείτε ότι ο λαό θα υπερψηφίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θεωρείτε είχατε προβλέψει ότι και σήμερα θα είστε παρόν. Εγώ θεωρώ ότι η κρυστάλλινη σφαίρα σα είναι λάθο. Προβλέπετε αν θα σα υπερψηφίσει η Επιτροπή να ε, γίνετε επίτροπος. Χάρη στη δική σας στήριξη, κύριε Γουλφ, είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή θα καταλήξει σε μια λογική απόφαση για το τι θα με κάνει. Είπα αυτό που είπα για το ότι η Ένωση το 2019 θα έχει 28 μέλη, γιατί είναι η ελπίδα μου, η προσδοκία μου, αλλά και η πεποίθησή μου. Πρώτα απ' όλα, ότι θα υπάρξει δημοψήφισμα που μάλλον το επιθυμείτε, αν και στη χώρα σας ε, προσπαθείτε να μειώσετε την πιθανότητα να διεξαχθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα γίνει δημοψήφισμα και ότι μετά τις συζητήσεις ε, που θα έχουν γίνει για μεταρρύθμιση κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχει μια σαφή επιλογή ο, ο λαός του Ηνωμένου Βασιλεία και είναι σαφής η πεποίθησή μου και την έχω εδώ και καιρό ότι εάν έχουν να επιλέξουν μεταξύ μια ισχυρή και μεταρρυθμισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και αποχώρηση από αυτήν, οι Βρετανοί εκλογεί θα παραμείνουν. Θα αποφασίσουν να παραμείνουν. Γι' αυτό είπα ότι αυτό πιστεύω ότι θα είναι η πραγματικότητα το 2019. Διότι όταν θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα, ο λαό της χώρα μου θα καταλάβει ότι μερικέ από αυτέ τι ιδέε που αναφέρονται ότι θα υπάρχει πρόσβαση ε, μια που αναφερθήκατε σε όνειρα και παραμύθια, ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στην ενιαία αγορά με τους όρους που θα θέλει το Ηνωμένο δεν είναι πολύ πιθανό. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν θα αρχίσει η συζήτηση, όταν ε, οι ψηφοφόροι, οι επιχειρήσεις μεγάλες και μικρές από τις οποίες εξαρτώνται οι εργαζόμενοι και των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται από την ενιαία αγορά, τότε θα ψηφίσουν να παραμείνουν. Ευχαριστώ κύριος Μπερνάρ Μονό από τους μη εγγεγραμμένους. Γεια σας κύριε Χίλ. το παραβίθι σε μια ευτυχισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα, δεν, θα, δεν θα υλοποιηθεί. Γιατί έχουμε και τους συστημικούς κινδύνους και τις εξωτερικές συνθήκες. Προτείνεται να πρόγραμμα τλοποιημένων δανείων για τις τράπεζες, το IBC. Επίσης προσδιορίσατε στις απαντήσεις ότι το πρώτο τριμήνο θα προτείνετε κάποια μέτρα για ενίσχυση αγορά στη τλοποίηση. Τελευταία φορά όμως που είχαμε τέτοια αγορά, ε, ολοκληρώθηκε το 2008 με μια τραγική παγκόσμια τραπεζική κρίση και μάλιστα τα δημόσια κονδύλια τόνωσαν τότε το ιδιωτικό ε, τραπεζικό σύστημα. Και από το 2008 μέχρι το 2011, 13% του ΑΕΠ δόθηκε σε άμεσες ενισχύσεις και ε, χρηματοπιστωτικές εγγύησεις. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνετε για να εναχαιτήσετε την κερδοσκοπία των ιδιωτών ε, επενδυτών και φορέων και τι μέτρα θα πάρετε σε περίπτωση παραβίασης αυτού του μηχανισμού ελέγχου που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπούμε που και εσείς ε, πιστεύετε ότι μία θετική πρόβλεψη και ένα θετικό όραμα για το μέλλον είναι μόνο παραμύθι, είναι ένα απλό παραμύθι. Και πιστεύω ότι θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εργαστούμε και με σωστή προσπάθεια όλα είναι δυνατά. Σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση, θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ της τιτλοποίησης υψηλής ποιότητας και της πιο επισφαλούς ή επικίνδυνης τιτλοποίησης. Συμφωνώ ότι κανένας δεν θέλει να παλινδρομήσουμε και να επανέλθουμε στους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Και νομίζω όμως ότι υπάρχει μια αυξανόμενη συνένεση ότι είναι δυνατόν να αποκομίσουμε καρπούς και πλονεκτήματα από, μια, από ασφαλή μέσα τιτλοποίησης. Και αν δεν κάνω λάθος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο ζήτησε τη θέσπιση ενός γενικού ρυθμιστικού πλαισίου και τον ορισμό τιτλοποίησης υψηλής ποιότητας. Νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε τέτοια μέτρα, αρκεί να είναι απλά και διαφανή, με μια σωστή στάθμιση των διαφόρων συμφερόντων. Και στις καταξιδότηση πράξη για τη δεύτερη αφαιρεγγιότητα και για τη ρευστότητα, θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση των διαφόρων επιπέδων τιτλοποίησης και μέσω τιτλοποίησης. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να προωθήσουμε και να είμαστε αισιόδοξοι. Να μην είμαστε ρηψοκίνδυνοι, αλλά ούτε να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες να ξαναπροσελκύσουμε παιδείς προς την οικονοματία. Ο κύριος Φούλβιο Μαρτουσέλο από το ΕΛΚ. Εγώ, κύριε Επίτροπε, δεν θα σας συγχαρώ και αν έχουμε συμπληρωματική ακρόαση είναι γιατί δεν μας είχατε πείσει στην αρχική σας ακρόαση. Έχω μια ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για τα stress test, αυτά τα τεστ αντοχής για τις τράπεζες που θα οργανώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι γνώμη έχετε για, τα, για την επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων. Είχαμε ήδη προβλέψει ότι πολλές τράπεζες δεν θα δώσουν με επιτυχία αυτές τις εξετάσεις αντοχής. Ποια είναι η γνώμη σας καταρχήν για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος. Και πιστεύετε ότι θα αναζωπυρώσετε την αγορά με την εξαγγελία τέτοιων κακών μαντάτων. Στο, ο αγγλικός τύπος σας χαρακτήρισε ευρωσκεπτικιστή. Ενώ εδώ μας δίνεται την εντύπωση φιλοευρωπαίου και θερμού ευρωπαϊστή. Μήπως ε, η υποψηφιότητά σας για τη θέση του Επιτρόπου επηρέασε τη συμπεριφορά σας. Καταρχήν, ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Η πείρα μου με δίδαξε ότι ο τρόπος που παρουσιάζει ο τύπος τους ανθρώπους και παντού, αλλά ιδιαίτερα στην ε, Μεγάλη Βρετανία, είναι ε, πολύ ρητός και κατηγορηματικός και μερικές φορές ομός, αλλά πολλές φορές άσχετος με την πραγματικότητα. Βρίσκομαι εδώ γιατί ενδιαφέρομαι για αυτή τη δουλειά και θέλω να διαδραματίσω το ρόλο που θα μου επιτρέψουν οι αρμοδιότητές μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τεστ αντοχής, ε, σίγουρα θα είναι δύσκολες αυτές οι εξετάσεις για τις τράπεζες και εσκεμένα γίνεται κάτι τέτοιο και μάλιστα μετά την πρώτη, τον πρώτο γύρο έγιναν πιο αυστηρά αυτά τα τεστ. Και ήταν πολύ θετική και η ανταπόκριση της αγοράς και οι θεσμικοί επενδυτές στη μεγάλη τους πλειοψηφία εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη διεξαγωγή αυτών των τεστ αντοχής. Θα ήταν πρόωρο και ανεύθυνο εκ μέρους μου να προεξοφλήσω, να προδικάσω τα αποτελέσματα αυτών των τεστ αντοχής. Θα δημοσιευθούν αργότερα τον Οκτώβριο. Οπότε και θα συμβούλευα και τους υπόλοιπους να αποφύγουν τέτοιες προβλέψεις. Να αφήσουμε τα αποτελέσματα να μιλήσουν από μόνα τους όταν δημοσιευθούν. Ήδη πάντως ε, γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες έχουν αυξήσει το ποιοτικό τους κεφάλαιο και είναι πάνω από 500 δισεκατομμύρια πια από το 2007 και πέρσι τον Ιούλιο είχαν κεφάλαιο πάνω από 140 δισεκατομμύρια ε, ε, κάνοντας την προετοιμασία για τα τεστ αντοχής. Οπότε παίρνω σοβαρά τα πράγματα, δεν θα, έχουμε καμία, δεν θα δείξουμε καμία επίοικια η συγκαταβατικότητα και θα φροντίσω μαζί με τους ε, συναδέλφους όλα τα μέτρα των ε, εποπτικών αρχών να τηρούν την ενωσιακή νομοθεσία και φυσικά και τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση που χρειαστούν δημόσια κονδύλια. Πάντως είναι καλά τα τεστ αυστηρά και δεν θα πρέπει από τώρα να κάνουμε προβλέψεις για την έκβασή τους. Υπερβάν από τους σοσιαλιστές. Κύριε Χίλ, αν είχα κάποια αμφιβολία για την εθνικότητά σας, ακούγοντας το είδος του χιούμορ σας, δεν έχω πια καμιά αμφιβολία. Οι απαντήσεις σας στα έγγραφα ερωτήματα, σε ό,τι αφορά την τίτλοποίηση, ανέφεραν ότι η πύλη θα πρέπει να μείνει Κλειστή σε πολύπλοκα διαφανή και επικίνδυνα χρηματοπιστωτικά μέσα. Μα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι και να ξεκινήσουμε και πάλι από την αρχή τη διαδικασία τιτλοποίησης και να μπορέσουμε να εμποδίσουμε τους κινδύνους να αναδυθούν οι οποίοι οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση που είμαστε ακόμα μέσα σε αυτή την κρίση και που οδήγησαν σε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη και σε ένα άκρατο κερδοσκοπισμό και τη δημιουργία φυσαλίδων. Ποιο είναι ο χρυσό κανόνα με τον οποίο θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε την καλή τιτλοποίηση από την κακιά. Πιστεύω <clears throat> ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι δεν μπορώ να διεκδικήσω την κατοχή ενός χρυσού κανόνος. Είναι πολύπλοκος ο χώρος και θα πρέπει να κάνουμε μια σειρά από κρίσεις, να Υπάρχουν μια σειρά αποφάσει από κοινού. Όταν δούμε παραδείγματο χάρη της κατεξουσιώσει πράξη για το Solvency 2 και επίση του κανόνε ρευστότητος των πιστοτικών ιδρυμάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξασφαλίσουμε με συνεργασία μεταξύ μα. Νομίζω ότι οι αρχέ που πρέπει να ακολουθήσουμε, που διαφέρουν φυσικά από ένα χρυσό κανόνα, αυτό το αναγνωρίζω, η αρχή πρέπει να ακολουθήσουμε είναι ότι η κλίδα για μια αγορά ε, τιτλοποίησης που είναι ασφαλής είναι η απλότητα και η κοινότης συμφερόντων. Να μπορούν να ξέρουν οι καταναλωτές τι είναι αυτά τα εργαλεία και πώς έχουν συσκευαστεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι απαραίτητη η διαφάνεια ώστε να μπορούν οι επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε δημόσια γνωστοποιημένες πληροφορίες και να μπορούν να κάνουν μια σωστή αξιολόγηση κινδύνων και πιστοτικών κινδύνων και επίσης ταυτότητα ή τουλάχιστον προσέγγιση συμφερόντων, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι εκδίδουν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο θα πρέπει να έχουν και οι ίδιοι μια συμμετοχή σε αυτό, ώστε να έχουν κάθε κίνητρο για να είναι ασφαλέ το εργαλείο αυτό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να καθοδηγηθούμε από αυτέ τι αρχέ. Πιστεύω ότι όπω είπα προηγουμένω θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο μαζί με του συναδέλφου από την Επιτροπή σας νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τιτλοποίηση υψηλή ποιότητα επί τη βάση των τριών αυτών αρχών που ανέφερα προηγουμένως και μια από τις πρώτες προτεραιότητες μου, αν εγκριθώ ως Επίτροπος, θα είναι να ξεκινήσω το παρασκευαστικό έργο για να υπάρξει αξιολόγηση του αντικτύπου μιας πιθανής πρωτοβουλίας στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Χούμπνερ, Τανούτα Χούμπνερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λόρδε Χίλ. Είσαστε αυτή τη στιγμή υποψήφιος για να αναλάβετε ένα κλάδο που είναι ιδιαίτερα δυναμικός. Ξέρουμε ότι συνέχεια έρχονται στην επιφάνεια νέα εργαλεία στο χρηματοπιστωτικό τομέα και αυτό ξεπερνάει πολλέ φορέ την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει τα θέματα αυτά. Ένα τρόπο για να τα αντιμετωπίσουμε αυτά, όπω είπατε, είναι το να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που μα δίνουν κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ενώ αντί να περάσουμε άλλα δύο χρόνια για να τροποποιήσουμε του κανονισμού. Για να επιτύχει όμω αυτό χρειάζεται μια καλή συνεργασία που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τη Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμεί σημειώσαμε ότι η Κομισιόν μερικέ φορέ φορές διστάζει να λάβει υπόψη την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν επεξεργάζεται τις ε, ε, πράξεις αυτές, όπως παραγωγός χάρη για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό ε, και τον ενιαίο μηχανισμό επίλυσης. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε εσείς να εξασφαλίσετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι θεμητές του ανησυχίες θα λαμβάνουν υπόψη από την Κομισιόν και θα έχουμε το, την ικανότητα να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τις κατάλληλες λύσεις μέσω της διαδικασίας αυτής χωρίς καθυστερήσεις. Πρώτα απ' όλα, για την αρχή της ε, ερώτησής σας, συμφωνώ μαζί σας. Είναι πάρα πολύ δυναμικός ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και θα πρέπει να παραμείνουμε ενήμεροι για όλες αυτές τις εξελίξεις, όπως ακριβώς είπατε, η κατεξουσιοδότηση πράξης είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη αυτή ταχύτητος, γιατί μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα με την νομοθεσία επίπεδου 1 και μας δίνει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε για να, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις πράξεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κανονισμούς ή οδηγίες. Συμφωνώ μαζί σας, προφανώς, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα κέριο ρόλο εδώ, γιατί πρόκειται για νομοθεσία επίπεδου 1, αυτή είναι η νομοθεσία η οποία δίνει τις εντολές της Κομισιόν για να εκδώσει νομοθεσία επίπεδου 2, κατεξιοδότηση δηλαδή, πράξεις. Εδώ είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σαν νομοθέτη που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχει και το δικαίωμα να αντιταχθεί σε νομοθεσία επίπεδου 2 ως Κοινοβούλιο. Σίγουρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε όλα αυτά, όπως λέει και το δεύτερο σας ερώτημα. Η δική μου δέσμευση απέναντί σας είναι ότι θα εργαστώ σε ένα πνεύμα συνεργασία που Πιστεύω ότι αυτό ήταν που ανέπτυξε και ο προκάτοχός μου κύριος Μπαρνιέ και θα προσπαθήσω να σταθώ και εγώ στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή είναι λοιπόν η δέσμευση που μπορώ να σας δώσω. Σε γενικές γραμμές όμως, νομίζω ότι σε αυτό το τομέα που είναι ρευστός και εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρενάτο Σόρου από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Χίλ, όταν περιγράψατε προηγουμένω. Ε, τι θα γίνει την επόμενη πενταετία. Αναφερθήκατε στο 2019 στην έννοια αγορά κεφαλαίων που θα αντιδρά σύντομα, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας για μια έννοια αγορά κεφαλαίων λοιπόν η οποία θα ήταν επίσης προσεκτική, δεν θα ε, ήταν ιδιαίτερα κίνδυνη. τις επόμενες εβδομάδες. Το Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, θα ασχοληθεί με κείμενα που αφορούν την ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα μιλήσουμε πολύ για την ανάγκη της διαφάνειας. Γιατί ξέρετε ότι αυτή η αγορά είναι τεράστια εν δυνάμει, 535 δις. Είναι διπλάσια από την Αμερικανική και επταπλάσια από την Κινέζικη ε, ανάλογη αγορά. Ε, μια που μιλάτε για διαφάνεια, μήπως ε, δεν πρέπει να καθορίσουμε κάποια όρια για να αποφύγουμε μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση που θα ήταν τρομερά οδυνηρή. Νομίζω ότι η βασική ερώτηση που θέσατε για την ε, σημασία της διαφάνειας με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Φυσικά χρειαζόμαστε διαφάνεια σε όλες μας τις ενέργειες ε, ρύθμιση της αγοράς. Οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι επενδυτές όταν αγοράζουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα είτε είναι ε, υποθήκη, είτε είναι μετοχή, είτε είναι ασφάλεια. Πρέπει να ξέρουν ε, ποιες είναι οι κρυφές πλευρές του κόστους. Πρέπει όλοι οι επενδυτές να γνωρίζουν σε τι επενδύουν. Και γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη σωστής τιτλοποίησης, όπως το έθεσε προηγουμένως και η κυρία Μπερέζ. Χρειάζεται επίσης διαφάνεια. Για παράδειγμα, αν θέλει να αναπτύξει κανείς μια αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επενδύουν οι μικρομεσαίες, και όλοι νομίζω το επιθυμούμε, οι επενδυτές πρέπει να έχουν τη σωστή ενημέρωση για το πώς λειτουργούν, τι είναι αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου εύκολη πρόσβαση σε αυτή την ενημέρωση, υπάρχει πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός της αγοράς. Το βασικό λοιπόν σημείο που προσπαθείτε να τονίσετε περί διαφάνειας είναι απόλυτα ορθό και θα επιδιώξουμε να υπάρχει σε όλες μας τις ενέργειες. Είτε, είτε έχει να κάνει με ρυθμίσεις, είτε με καταναλωτικά προϊόντα, είτε με οποιοδήποτε κανονισμό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κάρας από το ΕΛΚ. Κύριε Χίλ, καλώς ήρθατε. Να πω κάτι για την εισαγωγική σας ε, παρέμβαση. Έχω μια σαφή ερώτηση. Μας ε, δώσατε πολλές ωραίες εικόνες. Ποιες είναι οι τρεις κυριότερες προτεραιότητές σας, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό το όραμα που δημιουργήσατε. Και από αυτές τις τρεις συγκεκριμένες προτεραιότητες, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ποιο είναι το πρώτο στοχευμένο μέτρο και πού θεωρείτε ότι θα είναι οι αδυναμίες των προσπαθειών σας. Ε, είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει κανεί μόνο τρει ε, γιατί στην εισαγωγική μου ομιλία αναφέρθηκα σε πέντε. Οι τρεις ε, που πιστεύω ότι και από πλευρά ε, έμφυτη σταθερότητα του συστήματο και από πλευρά εργασία πρέπει να γίνει τώρα, θα μπορούσαν να είναι. Είναι ολοκλήρωση τη εργασία ε, για να προωθηθεί η Τραπεζική Ένωση. Εδώ πρέπει αμέσως να αναλάβουμε ενέργειες. Τώρα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που ήδη έχουν, είναι εν εξελίξη. Το δεύτερο θα ήταν η Ένωση Κεφαλαιαγορών και για τα πρώτα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση έχω ήδη μιλήσει. Έχω πει σε ποια θέματα θα μπορούσαμε αμέσως να έχουμε πρόοδο στο ELTIF, στην αγορά για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων, πώς θα ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις των μικροεπενδυτών. Η Κομισιόν έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για αυτά. Αυτό ήταν ο δεύτερος τομέας μου. Και ο τρίτος τομέας είναι κάτι το οριζόντιο θα έλεγα για τις μικρομεσαίες γιατί θεωρώ ότι αν μπορέσουμε να λάβουμε μια σειρά από μέτρα, ορισμένα ήδη τα ανέφερα, αλλά θα υπάρξουν και άλλα, η οδηγία για τον εμπνευματικό φυλάδιο για παράδειγμα, εάν μπορούμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό νομίζω και στην ερώτησή σας να είναι στοχευμένες πάντα οι προσπάθειές μας αυτό νομίζω είναι ζωτική σημασία οποιαδήποτε επιχείρηση οποιοδήποτε τραπεζικός οργανισμός οποιαδήποτε, οποιοδήποτε υπουργείο μπορούν να επιτύχουν αν οι ενέργειες είναι στοχευμένες έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο οπότε ο τρίτος τομέας για μένα θα ήταν τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες Σας ευχαριστώ Σαν ποτέρχο από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας, Λόρδε Χίλ. Την περασμένη φορά μία από τις ερωτήσεις μας ε, αφορούσε την ε, ισοδυναμία της τρίτης χώρας της σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, παρόμοιες προκλήσεις θεωρείται ότι θα έχουμε και σε σε διαπραγματεύσει με άλλε χώρες και περιοχές του κόσμου. Νομίζω ότι το... μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι εστιαζόμαστε αποκλειστικά στη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. και πολύ σωστά επισημάνατε και πολύ σωστά μα υπενθυμίσατε ότι έχουμε ζωτικά συμφέροντα και σε άλλες περιοχές του κόσμου και με άλλες χώρες. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με αυτό τον επενημό και την υπενθύμηση, γιατί έχουμε και ε, χρηματοπιστωτικά κέντρα στην Ασία, στο Χονγκ Κόνγκ, δηλαδή και τη Σιγκαπούρη, ε, που αναπτύσσονται ραγδαία, οπότε δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες ε, και τη ραγδαία εξέλιξη των συγκεκριμένων κλάδων στην Ασία, για παράδειγμα. Και για να λάβουμε και αυτό το θέμα υπόψη, όπω είπαμε και πριν με, την κυρία Γκουλάρ, θα πρέπει να έχουμε ισχυρού κανόνες για την τρίτη χώρα για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος προς το συμφέρον των καταναλωτών και έχουμε, θέλουμε και μια συντονισμένη ε, ρυθμιστική μεταρρύθμιση. Και στην προσέγγιση μας ε, θα φροντίσουμε ώστε και τα αντίστοιχα μέτρα των άλλων ε, χωρών να είναι ισοδύναμα με τα δικά μας. Έτσι θα έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία των παγκόσμιων αγορών. Και σε καμία περίπτωση θα πρέπει να χάσουμε τη φόρα μας σε αυτή την προσπάθεια και να αποφύγουμε ασυνεπή ή ε, ευαλωματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, κάτι που θα μας οδηγήσει στη διαιτησία. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και τους δεσμούς μας με τις αναδυόμενες οικονομίες και τις αναδυόμενες αυτές ε, αγορές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο G20 και στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ε, θα θέσει το θέμα των διαδικασιών ε, εξασφάλισης αντιστοιχείας ισοδυναμίας. Και θα σας ενημερώνω για την πρόοδο που θα σημειώνουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές, ζητώντας και τη δική σας άποψη. Πάντως ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα από τους φιλελεύθερους Βαρχόιζεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, εδώ είμαι κύριε Χίλ. Σας ευχαριστώ για τις ε, γραπτές απαντήσεις που στείλατε στις ερωτήσεις μας για την ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Πολύ διεξοδικές οι απαντήσεις. Για παράδειγμα, λέτε στις απαντήσεις σας ότι μερικά εμπόδια είναι ήδη γνωστά για την ολοκλήρωση αυτής της Ένωσης αγορών. Τι εννοείτε, γιατί είπατε ότι οι προτεραιότητες μου για έγκαιρη δράση είναι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εμπόδια εκεί που είναι σαφή τα προβλήματα και οι λύσεις είναι ε, εμφανείς πια. Και δίνετε τρία παραδείγματα. Προδιαγραφές για υψηλής ποιότητας τυπλοποίηση, κοινά αξιόπιστα πρότυπα για πρόσβαση των καμεσών επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση και διευκόλυνση της, ε, η ανάπτυξη αγοράς για την ιδιωτική τοποθέτηση. Πολύ, πολλά υποσχόμενα όλα αυτά και η ερώτησή μου είναι πώς ορίζεται την έγκαιρη δράση ή της, α, την άμεση δράση που υποσχεθήκατε. Πότε να περιμένουμε δηλαδή συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν ξέρω αν και στη δικιά σας χώρα έχετε μία παρόμοια, πα... μία παρόμοια εκφρασία. Όταν λέτε ότι κάτι επίκειται, λέτε αναμένεται για την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και συνήθως ε, γίνεται κάτι τέτοιο το χειμώνα. Αυτό δεν θα συμβεί όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν το θέμα είναι κέριο. Ε, έχει νευραλική σημασία και θα πρέπει να το βάλουμε στις ράγες το συντομότερο δυνατό. Και μία από τις προκλήσεις μας είναι να δημιουργήσουμε αυτή την όθηση, τη φόρα και φυσικά ε, θέλουμε να εμπλέξουμε και τις 28 χώρες μέλη για να σημειώσουμε πρόοδο. Εγώ είμαι υπέρ της ε, ταχείας πρόοδου. Και μπορεί την περασμένη εβδομάδα να έδωσα την εντύπωση ότι κολλήσει αργό κάπως, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα φροντίσω να γίνουν ε, διεξοδικές οικονομικές αναλύσεις, εμπεριστατωμένες για τα διάφορα θέματα, τα εμπόδια και τον τρόπο υπέρβασης τους. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε και θα το ξεκινήσω πάραυτα από την πρώτη μέρα και όλα ανάληψης των καθηκόντων μου, αν εγκρίνεται φυσικά. Και φυσικά θα σας ενημερώσω και θα υποβάλω προτάσεις, θα έχουμε συγκεκριμένες διαβουλεύσεις και διεξοδικά προγράμματα δράση. ώστε να τα συζητήσουμε, να τα αποφασίσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Επιπλέον, ορισμένα πράγματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Ε, αγορά, ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΕΛΤΙΦ, ε, ε, ιδιωτική τοποθέτηση, όλα αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Οπότε εκεί θα πρέπει να αφήσουμε αμύωτη την πίεση και την προσπάθεια και να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο πάρα αυτά, το συντομότερο δυνατό. Το θέμα επήγει και πιστεύω ότι όλοι συμμεριζόμαστε την επιτακτική ανάγκη α, ανάληψης δράσης. Ευχαριστώ κύριος Πέτερ Σάιμον. Κύριε υποψήφιε Χιλ, ε, Επιτροπέ Χιλ, στις ε, απαντήσεις σας μέχρι τώρα έχετε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μακροχρόνια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, όμως είναι όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικέ οι προτάσεις σας για τη δημιουργία μιας κοινής, ενός κοινού συνόλου κανόνων για τις ε, αποταμίευσεις. Πολλοί φοβούνται ότι θα μπορέσει με τον τρόπο αυτό να αποδυναμωθεί η ουσιαστική λειτουργία των ε, τραπεζών και επομένως χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς αντιμετωπίζετε την ιδέα του να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συνεχίσετε αυτή την πρόταση του Μισελ Μπαρνιά. Ένα δεύτερο ερώτημα για τα θέματα της ε, του διοικητικού άχθους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Λέτε ότι η μείωση του άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Στο τελευταίο, στην τελευταία θητεία χρειάστηκε όμως να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες, χρειάστηκε να υπενθυμίσουμε στην Κομισιόν ότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό έχει να κάνει και με το μηχανισμό επίλυσης. Ελπίζω ότι αυτό θα θεωρηθεί πλέον ότι είναι κάτι το προφανές. Το δέχεστε εσείς αυτό ότι είναι κάτι το αυτονόητο. Καταρχήν, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη σε επιχειρήσεις και φυσικά και σε τραπεζικά ιδρύματα και είναι απαραίτητο να το αναγνωρίσει κανείς αυτό και θα πρέπει να έχουμε μια λογική διαφοροποίηση στα θέματα αυτά. Είτε πρόκειται για την ενθάρρυνση της τιτλοποίησης, για να έχουμε τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας, είτε μιλάμε για το ρυθμιστικό άχθος για τις μικρές επιχειρήσεις ή να μην έχουμε μια προσέγγιση που δεν κάνει διάκριση μεγέθους στις επιχειρήσεις, είτε όταν μιλάμε για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να θεσπιστούν για να κάνουμε ασφαλέστερο το τραπεζικό μας σύστημα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές ιδιαιτερότητες και τις επιπτώσεις του μεγέθους για τα πιστοτικά ιδρύματα. του. λεχθέντος, όταν πρόκειται για την συμμετοχή που θα πρέπει να κάνουν οι διάφορες τράπεζες στο Ταμείο Εξυγίανσης ή σε άλλους ε, φορείς, αυτό είναι κάτι το οποίο ωφελεί όλες τις τράπεζες και θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως το οποίο αναφέρεται η κυρία Σίμων για τη διαφοροποίηση νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοφροσύνη και ευφυΐα σε όλους τους χώρους και αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε απρόσεκτοι ή ότι θα, παίρνουμε, θα κάνουμε μονάχα βολονταριστικές αποφάσεις για την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών θεμάτων θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευφύς σε σχέση με την εκτίμηση διαφόρων επίπεδων κινδύνου. Σε σχέση με το πρώτο σας ερώτημα, Νομίζω ότι η απάντησή μου θα ήταν ότι σε σχέση με τις επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ένωση Αγορών, στην μελλοντική αυτή αγορά, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα και θα σας έλεγα, και αυτό είναι βέβαια μια ιδέα που εσείς υποστηρίζετε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να το συζητήσω μαζί σας, μπορούμε πράγματι να διερευνήσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες ή ποιες είναι οι δυσκολίες που συνάπτονται με μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ. Ζητώ από τους συναδέλφους να μένουν μέσα στο περιθώριο του χρόνου τους. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο για την απάντηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρία σε εγκαίρος. Ο Brian Hayes έχει το λόγο τώρα από το ΕΛΚ. Λόρδε Χιλ, καλώς ήλθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Κάποιοι συνάδελφοί μου φαίνεται να έχουν δυσκολίες ε, όταν εσείς κοιτάξατε την κρυστάλλινη σφαίρα σας και είδατε ότι το, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέμενε πλήρως προσιλωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019. Είναι πάρα πολύ καλό που ακούμε με τέτοιους σαφείς όρους ένα εξέχοντα Βρετανό πολιτικό να λέει κάτι τέτοιο. Γιατί οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ λοιπόν καθυσχαστικό αυτό το οποίο ακούμε. Εν ώψη αυτού κιόλας θα ήθελα να πω, να θέσω το εξή ερώτημα. Αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν ανησυχίες μεταξύ ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης, ότι ως Βρετανός Επίτροπος που έρχεσαι από μια ζώνη, από μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωζώνη, αλλά έχει την ευθύνη περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωζώνης, ότι αυτό μπορεί να είναι ένα επίμαχο θέμα. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο αυτό θέμα και πώς θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε, να παροτρύνετε μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρωζώνης παρά το γεγονός ότι εσείς δεν προερχέστε από μια χώρα της Ευρωζώνης πιστεύω, λέει ο κύριο ο Λόρδος Χιλ, πρώτα απ' όλα ότι το θέμα της ε, εργασίας που θα πρέπει να γίνει για να επιληθούν οι διαφορές ή να υπάρξει καλύτερη κατανόηση μεταξύ αυτών που συμμετέχουν και αυτών που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εγχειρήματο που θα πρέπει να υπομισθώ, ιδίω στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης. Και βλέποντας τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία από αυτή που είχε να αναλάβει ο Μισελ Μπαρνιέ όταν ήταν αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα αυτά. Υπήρχαν κάποιες δυσφορίες από χώρε οι οποίες δεν ήταν μέσα στη ζώνη του ευρώ, αλλά αυτά τα οποία έπραξε τα τελευταία πέντε χρόνια έδειξε ότι παρόλα αυτά μπορεί να λειτουργήσει ως επίτροπος κάποιος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις απόψεις μου για την Ευρωζώνη, νομίζω ότι πολύ σαφώς τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταδείξει ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση δεν ήταν επαρκής και δεν ήταν πλήρες το ευρωπαϊκό εγχείρημα ολοκλήρωσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για καλύτερη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, οι κανόνες του 6 ε, Pack και του 2 Pack και φυσικά και η Τραπεζική Ένωση που θα είναι στο χαρτοφυλακείο μου. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι κανόνε θα λειτουργήσουν στην πράξη και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να βελτιωθούν ή να συμπληρωθούν σε ορισμένε περιπτώσει. Ενδεχομένω η μακροχρόνια ενίσχυση και σταθεροποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί περαιτέρω ολοκλήρωση. Και η απάντηση στο ερώτημά σα λοιπόν είναι αν παρουσιαστούν στοιχεία που να δείχνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω ολοκλήρωση σε τομεί υπό την ευθύνη μου, εγώ σίγουρα θα έκανα μια πρόταση που να λαμβάνει υπόψη αυτό το γεγονός και είναι ορθό να πω ότι αντί να κοιτάω μια κρυστάλλινη σφαίρα για το μέλλον, κοίταζα μια κρυστάλλινη σφαίρα για το παρελθόν και ήμουν ενώπιον σας το 2012. Ελπίζω ότι τότε θα είχα μπορέσει να ε, προτείνω δράσεις όπως η Τραπεζική Ένωση και θα υποστήριζα τη δράση που έλαβε στη συνέχεια η Κομισιόν για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Μιγέλ Βιέγας από την ΚΟΕ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Δεν θεωρείτε ότι η πρόσβαση των επενδυτικών ταμείων στο μηχανισμό διακανονισμού των διαφορών ε, ε, μπορεί να επηρεάσει το θέμα της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και να δημιουργήσει προβλήματα στο θέμα αυτό. Τι γίνεται με την οδηγία 17 του 2014 που υποδίζει τις τράπεζες να ζητήσουν περαιτέρω πιστώσεις ε, μετά την ε, εκτέλεση της υποθήκης. Γιατί υπάρχει κάτι αντίστοιχο στις Ηνωμένες Πολιτείες και κρεμούν πολλές ε, δικαστικές αποφάσεις ως προς το θέμα αυτό. Θα κάνετε πιο φιλόδοξη την οδηγία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό διαχωρισμό. Συμφωνείτε με την πρόταση του κυρίου Λικάνεν που είναι υπέρ του πλήρους διαχωρισμού μεταξύ των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων και των κανονικών τραπεζικών εργασιών. Ή είστε υπέρ της αντιπρότασης του προκατόχου σας Μπαρνιέ που προτείνει μια διαφορετική λύση που στην ουσία καταλήγει στα ίδια αποτελέσματα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν κατάλαβα το τελευταίο σημείο σας. Ε, ίσως πρέπει να ε, συνεχίσω παρόλα αυτά και ε, εκτός αν ο πρόεδρος επιτρέψει να διευκρινίσετε. Παρακαλώ, ε, παραλαμβάνετε την τελευταία σας ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση για τον τραπεζικό διαχωρισμό. Είστε υπέρ του πλήρους διαχωρισμού των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων ε, από τις κλασικές τραπεζικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν την οικονομία. Είστε υπέρ μιας ενδιάμεση λύσης σαν αυτή που πρότεινε ο κ. Μπαρνιέ που επιτρέπει στις περισσότερες τράπεζες να περιορίσουν τις δραστηριότητες αλλά στο εσωτερικό μιας τράπεζας. Για το τελευταίο που αναφέρατε. Είχα την δυνατότητα ε, χοντρικά να κοιτάξω την ε, πρόταση που είναι συνέπεια των ποτάσεων Λίκανεν για το θέμα του διαχωρισμού των τραπεζών. Πώς θα αντιμετωπίζουμε το θέμα κάποιων τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν. Πρέπει όμως να εργαστούμε παραπάνω, περισσότερο από αυτού. Αυτά που έγιναν για την εποπτεία και για την εξυγίανση είναι σημαντικά αλλά για μερικές λίγες πολύ μεγάλες και πολύ περίπλοκες τράπεζες πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Από ό,τι έχω διαπιστώσει μέχρι τώρα υποστηρίζω την ε, ε, καλή πρόταση, ε, αντικειμενική πρόταση του κυρίου Μπαρνιέ. Ξέρω ότι ορισμένοι εδώ πιστεύουν ότι ε, δεν πηγαίνει αρκετά μακριά, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι υπερβολική. Άρα πρέπει να τα συζητήσουμε. Να δούμε πώ θα καταλήξουμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τραπεζών που είναι πολύ μεγάλε για να πτωχεύσουν και ίσω και άλλων ε, ιδρυμάτων. Πρέπει να μην εφησυχάζουμε και για άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εντός της Ένωσης και παγκοσμίως. Ε, Πολύ δουλειά. Τώρα για αυτό που είπατε για την συμφωνία TTIP και το ISDS. Όπως είπατε κι εσείς, είναι θέμα της συναδέλφου Σεσίλια Μάλστρομ. Εκείνη είναι αρμόδια και ξέρω ότι στην ακρόαση της είπε ότι είναι ακόμη υπερβολικά νωρίς για να πούμε ε, αν θα συμπεριληφθεί ο μηχανισμός διαιτησίας για τις διαφωνίες επενδυτών και κρατών στα πλαίσια των ε, διαπραγματεύσεων TTIP. Αλλά αν πρόκειται να συμπεριληφθεί, τότε είναι οπωσδήποτε σημαντικό να υπάρχουν και οι προληπτικές διατάξεις που συμπεριλήφθηκαν στις διαπραγματεύσεις ε, Ένωσης Καναδά. Ε, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ε, θα το συζητήσουμε μετά κάτι Για να απαντήσω στην μεσαία ερώτησή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μόρις Κοτ Κέιτο από τους Πράσινους. Μετά την προηγούμενη συζήτησή μας έχω ακόμη κάποιες αμφιβολίες για τη στάση σας έναντι της Ένωσης, αλλά η κύρια επιφύλαξή μου αφορά την ανεξαρτησία σας. Ακόμη και κάποιοι που σας στηρίζουν, που θεωρούν ότι ήταν σόφρον ο Γιούνκερ που σας έδωσε αυτό το χαρτοφυλάκιο, θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος να καθησυχάσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και για να μην έχουμε πολύ έντονες ε, διαμάχες με διάφορα συμφέροντα στην ε, Ένωση από τη μία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό για να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα σύγκρουση συμφερόντων, σα ρώτησα ε, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Για παράδειγμα το θέμα των ε, των τραπεζιτών και κάτι άλλο που σχετίζεται με αυτό. Πόσες φορές έχετε συναντηθεί επισήμως ή ανεπισήμως με τους David Cameron και George Osborne, πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών. Με ενδιαφέρουν και οι συναντήσεις στα διάφορα εξοχικά σπίτια ε, και οι συναντήσεις με τους υπουργούς επισήμως. Με συγχωρείτε. Δεν είμαι τμήμα του κύκλου φίλων των Κάμερον και Όσμπορν που μένουν στο Chipping Norton. Εγώ ε, μένω πολύ ήσυχα στο Σόλσμπερι και ε, δεν έχω πολύ στενή σχέση με αυτούς τους ιδιαίτερα γκλαμουριάριδες τύπους. Τους έχω δει βέβαια επανειλημμένα το τελευταίο εξάμεινο. Αλλά δεν έχω ημερολόγιο. Αλλά ως ε, επικεφαλής της Βουλής των Λόρδων τον ε, έβλεπα τον Πρωθυπουργό δύο φορές τη μέρα. Επίσης, όπως ξέρετε, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τη βδομάδα και πολλές άλλες συναντήσεις έχω με τον Πρωθυπουργό. Οπότε φυσικά τους έχω δει πολύ συχνά τον τελευταίο 1,5 μήνα το διάστημα που είμαι επικεφαλής της Βουλής των Λόρθων. Τώρα για την ερώτηση που κάνατε, πώ αντιμετωπίζω αυτά τα θέματα, τα θέματα της ανεξαρτησία που είναι πολύ σημαντικά. Έχω δώσει ήδη μια απάντηση, δεν μπορώ παρά να την επαναλάβω. Και από πλευράς των ε, νομικών υποχρεώσεων, των ηθικών υποχρεώσεων μου, λόγω του ότι θα ορκιστώ και από πλευράς της προσωπικής μου ε, φιλοσοφίας που είναι πάντα η προσπάθεια ε, να είμαι ειλικρινής, να μην υπόσχομαι ότι δεν μπορώ να κάνω αλλά ότι πω να το κάνω θα συνεχίσω εάν με εγκρίνεται να εργάζομαι με αυτόν τον τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις και έχω μια απόλυτα σαφή υποχρέωση να συμπεριφέρομαι με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον όπως όλοι οι επίτροποι και θα είχατε κάθε απέτηση να φερθώ έτσι θα είχατε κάθε απέτηση να μου ζητήσετε να λογοδοτήσω αν όχι και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάτρικ Οφλίν, EFDD. Λόρδε Χίλ. Υπόθηκε αυτή την εβδομάδα ότι ο Λίντον Κρόσμπι που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού είπε ότι δεν θα πρότειναν κανένα βουλευτή για να μην υπάρξει πραγματική εκλογή. Μήπως θεωρείτε ότι γι' αυτό σας πρότειναν εσά, μια που δεν έχετε εκλεγεί και είστε Λόρδος. Και κάτι άλλο. Κάποιος ε, αρθρογράφος είπε ότι μπορεί να είστε εδώ λόγω του ερωτήματος ακριβώς ε, γιατί κάποιος που δεν είναι στην Τραπεζική Ένωση είναι δυνατόν να είναι επίτροπος για την Τραπεζική Ένωση. Μας λέτε συνέχεια ότι είστε υπέρ της πιο συχνής ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσατε. Με συγχωρείτε. Α, η πρώτη σας ερώτηση. Για την πρώτη σας ερώτηση. Γιατί ανέλαβα, γιατί μου πρόσφεραν αυτήν την θέση. Γιατί μου την πρόσφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό γιατί έκανε αυτή την πρόταση. Ε, με χαρά θα σας δεχτεί, ίσως στο Κλάκτον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ε, αναφορά στο ότι θα γίνει αναπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον. Γιατί αυτό μόλισε στο UKIP ο, ο συντηρητικός βουλευτής εκεί. Ε, βεβαίως, ε, όπως ξέρετε, Ήμουν υπουργό που ε, πέρασε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ε, παιδείας. Επίσης ε, στο δεύτερο νομοθετικό σώμα ως Λόρδος βοηθώ να περάσω νομοθεσία και επίσης ήμουν σύμβουλος. Εργάστηκα και στον επιχειρηματικό τομέα, άρα έχω ένα κράμα δεξιοτήτων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εδώ. Γιατί δέχτηκα την υποψηφιότητα. Επειδή θεώρησα ότι θα μπορούσα να συμβάλλω στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου στην παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι από αυτού διαφωνούμε. Αλλά γι' αυτό είπα ναι στην πρόταση που μου έγινε. Και πώς θα προσεγγίσω τα καθήκοντά μου και για όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε τώρα μικροπολιτικά παιχνίδια με το ότι θέλω να εργαστώ σοβαρά για την Ένωση σε μια κρίσιμη φάση Τη Ευρωπαϊκή και παγκόσμιας ιστορίας. Ναι, το επιθυμώ. Αυτό είναι το κίνητρο για το οποίο δέχτηκα την υποψηφιότητα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ. Είναι Η Ναγκίλα από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ. Λόρδα Χίλ. Έχω δύο σχόλια που ήδη καλύφθηκαν μέρη. Καταρχήν για τι ε, τράπεζες που παρά είναι μεγάλες για να καταρρεύσουν. Παρά την τραπεζική νομοθεσία, που έχουμε εγκρίνει, το μέγεθο και η περιπλοκότητα μερικών από τι μεγαλύτερε τράπεζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα. Και πέρυσι οι μεγαλύτερε τράπεζε του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβαν ε, έμεση ενίσχυση 38 δισεκατομμυρίων από τα χρήματα των φορολογουμένων. Πώς θα αποφύγουμε οποιαδήποτε έμεση ε, ενίσχυση από τους φορολογουμένους ε, και πώς θα εφαρμόσετε κάτι τέτοιο και μάλιστα μεσοπρόθεσμα, ε, σε ποιο χρονοδιάγραμμα μάλλον, σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση. Ρώτησαν και οι συνάδελφοι πώς, ε, πόσες φορές ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να μπει σε μια δέσμη και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μετατραπεί στην, στο διάβλο που θα περάσει από τα διάφορες πιστοτικές μορφές. Καταρχήν για τις too big to fail τράπεζες, πολύ μεγάλες τράπεζες, είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό αυτό το θέμα και φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Και οι πρωτοβουλίε του κυρίου Μπαρνιέ, του προκατόχου μου για την Τραπεζική Ένωση, πραγματικά δημιούργησαν αισθητή πρόοδο, ενίσχυσαν την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος, αλλά υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός πολύ μεγάλων τραπεζών με Τυχαία του ενεργητικού που περβαίνουν μερικές φορές και το ΑΕΠ, ε, ολόκληρο το ΑΕΠ μιας χώρας και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Πάντως, η πρόταση Λίκανεν για την περαιτέρω ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Επίσης, και το ε, Συμβούλιο Χρηματοπιστής Σταθερότητας ε, έλαβε υπόψη αυτό το θέμα τη ε, συνολικής ικανότητας απορρόφησης των ζημιών που θα πρέπει να την αναλαμβάνουν οι τράπεζες ενισχύοντας το κεφάλαιό τους. Φυσικά θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να εξετάσουμε κατά πόσο και σε άλλους τομεί υπερβολικά μεγάλα ιδρύματα χρήζουν κάποιες ρύθμισης και θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποια μέτρα για την τιτλοποίηση θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να ενθαρρύνουμε ασφαλή τιτλοποίηση. Και δίκιο έχετε ότι η πρόκλησή μας είναι να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Και γι' αυτό αναφέρθηκα στις τρεις ε, αρχές. Την ε, απλότητα, τη διαφάνεια και την ε, στάθμιση συμφερόντων. Νομίζω ότι με βάση αυτές τις αρχές θα θεσπίσουμε ένα πλαίσιο, θα πρέπει όμως να το αναλύσουμε πιο διεξοδικά. Ο κύριος Μπουρκχάρτ Μπάλτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λόρδε Χίλ, θα μιλήσω στα γερμανικά. Χαίρομαι για την παρουσία σας και πάλι σήμερα για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε την, τον διάλογο μας. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα για σας. Πρώτα απ' όλα, λέτε καταρχήν στις γραπτές σας ε, ε απαντήσεις ότι υποστήριζετε την αναλογικότητα και ότι είναι μια θεμελιώδης αρχή της ε, πρότασης, των προτάσεων της Κομισιόν. Μπορείτε να μας διαβεβαίωσετε ότι και στις κατεξουσιοδότηση πράξεις θα είναι κανόνας η αναλογικότητα και ως μελλοντικό επίτροπος θα εξασφαλίσετε ότι η, ο φορέας για τις ε, αγορές και τα ομόλογα καθώς και για τις επαγγελματικές ε, συντάξεις και τα άλλα θα παίξει αυτό το ρόλο στην αναλογικότητα. Επίσης, μπορούν, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα έχουν πρόσβαση και οι Ευρωπαίοι πολίτες στην ε, πρόσβαση σε κάθε είδους ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και εναλλακτικά. Πώς θα το εξασφαλίσετε αυτός ο Επίτροπος. Για τα θέματα των ε, συντάξεων και των συνταξιοδοτικών ταμείων, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προτάσεις που έχουν ήδη ε, αντιμετωπιστεί στον τομέα αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η επεξεργασία τους. Δεν πρέπει εμείς να αποθαρρύνουμε την αγορά συνταξιοδοτικών ταμείων. Θα ήταν καλό στην Ευρώπη να μπορούμε να έχουμε περισσότερη επένδυση στα συνταξιοδοτικά ταμεία, κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα λοιπόν να κάνω και σαν τμήμα της ε, Ένωσης Κεφαλαγορών, αλλά και από την οπτική γωνία των καταναλωτών είναι να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα πέρα και από τα εθνικά σύνορα για να βοηθήσουν τους ε, πολίτες μας να αντιμετωπίσουν τα γυρατιά γιατί έχουμε αυτή την πρόκληση ενός γυράσκοντος πληθυσμού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για την αναλογικότητα τώρα. Σε γενικές γραμμές εγώ υποστηρίζω ιδιαίτερα να ακολουθήσουμε το δρόμο της αναλογικότητας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μερικές, μερικούς από τους μικρότερους χρηματοπιστωτικούς φορείς δεν θίγονται από υπερβολικά βαρύ άχθος κανονισμών και ρυθμίσεων. Πολλές φορές μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι κανονισμοί, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαιο που αλλιώς δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και αυτή την πτυχή. Θα πρέπει να δούμε το, την οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο για να δούμε αν υπάρχει γνωστοποίηση στο επίπεδο που θα πρέπει να υπάρχει και επίσης όταν αποφασίσουμε τη συμβολή των τραπεζών στο Ταμείο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ειδικό βάρος των μικρών και των μεγάλων τραπεζών θα εξισορροπούνται με το σωστό τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και να είναι μια κέρια αρχή που ακολουθούμε πάντα και θέλω να συνεργαστώ και μαζί σας και με όλους τους άλλους για να δούμε πώς είναι η τομή όπου μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα αυτή η αρχή της αναλογικότητας. Ευχαριστώ η Κέιτ Σουίνμπορν. Σας ευχαριστώ Λόρδε Χίλ. Πριν από λίγο στην ερώτηση της ε, Νίνα Γκίλ, αναφερθήκατε στι τράπεζε που είναι too big to fail, πολύ μεγάλες για να στοχίσουν. Στην τελευταία μα θητεία περάσαμε μια νομοθετική ρύθμιση που ακολουθούσαμε του κανόνε των G20 να υπάρχει η υποχρεωτική, ε, ο υποχρεωτικό συμψηφισμό των αγορών ομολόγων μέσω κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Και αυτό παίζει κάποιο ρόλο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του too big to fail. Εσείς θα εξασφαλίσετε λοιπόν ότι οποιοδήποτε πλαίσιο που θα δημιουργήσετε για την ε, επίλυση και την ανάκτηση προστατεύει τα στοιχεία ενεργητικού των πελατών των τραπεζών αυτών. Σας είπα και σε ένα προηγούμενο ερώτημα απαντώντας προς την ε, κυρία Γκίλ όλο αυτό το πλέγμα των ερωτημάτων γύρω από το too big to fail μπορεί πράγματι να ξεπεράσει και το στενό τομέα των τραπεζών, το παράδειγμα το οποίο στο οποίο αναφερθήκατε των κεντρικών αντισυμβαλωμένων είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Χρειάζεται πράγματι να το εξετάσουμε. Τα μέτρα τα οποία <clears throat> έχουμε αναλάβει ε, στην οδηγία ΕΜΙΡ για την ε, χρηματοπιστωτική υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ότι εκτός αγορά συναλλαγές γίνονται με πιο σταθερή βάση, αλλά αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνουμε και το ρίσκο σε μια μικρή ομάδα ε, φορέων. Πιστεύω ότι η πιο σύντομη απάντηση στο ερώτημά σας και ίσως και η καλύτερη απάντηση είναι ότι η πρόθεσή μου ήδη από την πρωτοχρονιά να έρθω ενώπιον σας με μια πρόταση για την ε, επίλυση μη τραπεζικών φορέων που περιλαμβάνουμε και σε αυτούς και τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους επί τη βάση των γνωστών σε μασίδι κινδύνων και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πράγματι την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προστατεύσουμε τους ε, φορολογόμενους μας σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία των ε, διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού Προς το παρόν δεν μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να πω οτιδήποτε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει καταρχήν μια αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά το προπαρασκευαστικό έργο στο οποίο αναφέρθηκα ήδη έχει ξεκινήσει, πρέπει να συνεχιστεί και εν καιρό θα έρθω ενώπιον σας με μια πρόταση. Ευχαριστώ. Και τελευταίος μας ομιλητής, ο κύριος Πέτρ Γέζεκ. Ευχαριστώ. Μια και έχω το προνόμιο και την τιμή να είμαι ο τελευταίος ομιλητής, θα υποβάλω λιγότερο τεχνικές και πιο γενικές ερωτήσεις. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, παρόλο που δεν το είπατε στην γραπτή σας δήλωση, φαντάζομαι ότι ε, σας αρέσει να ε, ασχολείστε με την Κυπουρική. Οπότε, αν σας αρέσει όντως η Κυπουρική ε, τι φυτά θα, ε, θα φυτέψετε πρώτα και τι, τι, μέτρα θα θεσπίσετε για να ανθίσει το χαρτοφυλάκιό σας την επόμενη πενταετία. Ποια... Επίσης, ε, πώς αντιλαμβάνεστε τις ανησυχίες μας για το ρόλο σας ως Επιτρόπου στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας και πώς θα λάβετε υπόψη και θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ανησυχίε σε περίπτωση που επιβεβαιωθείτε ως Επιτρόπος. Το πρώτο σας σχόλιο. Δεν είμαι και πολύ καλός κυπουρός. Και σίγουρα δεν είναι αυτή η κατάλληλη εποχή για φύτεμα σπόρων, αλλά για κλάδεμα, για σκάψιμο. Νομίζω ότι το φθινόπωρο αυτές είναι και οι πολιτικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Επίσης, ε, αν εξετάσουμε την νομοθεσία και τη συζήτηση που είχαμε για την αναλογικότητα και προκειμένου να έχουμε ρευστές επενδύσεις, ε, υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση και προσέλκυση επενδύσεων, ίσως θα πρέπει και το κλάδεμά μας είναι πολύ προσεκτικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανθοφορία και τον προγραμματισμό για τη σπορά και το, τα φυτέματα που θα κάνουμε του χρόνου, φυσικά προτεραιότητά μας θα είναι η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Και θα πρέπει να φυτέψουμε από νωρίς, να βάλουμε από νωρίς τα φυτά στο έδαφος με πολύ λίπασμα, ώστε να έχουν ραγδαία ανάπτυξη. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι είναι κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή θα είναι η εμπειρία μου που θα προσφέρω από το χώρο των μικρομεσαίων. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν τα μεγάλα ιδρύματα, οι ρυθμιστικές αρχές ή τα κράτη ε, συμπεριφέρονται σαν να είναι όλες οι επιχειρήσεις ίδιου μεγέθους ε, αυτό ταλανίζει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, γιατί μπορεί οι μεγάλε επιχειρήσει να μπορούν να συμμορφωθούν με κάποιου κανόνες, αλλά δεν έχουν την ίδια πολυτέλεια και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και μερικέ φορέ με υπερβολική γραφειοκρατία αποκαρδιώνουμε του ε, νέου επιχειρηματίε να εισέλθουν στην αγορά. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Και σε ένα άλλο το με περιμένω καρποφορία είναι η Τραπεζική Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που άντλησα, νομίζω το πιο σημαντικό που έχω να ε, θυμηθώ και να λάβω υπόψη από τις ανησυχίες σας είναι η ανεξαρτησία. Γιατί είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε επανειλημμένως και στις συζητήσεις που είχα με πολλά μέλη της Επιτροπής. Σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την ανεξαρτησία μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω παρά να δηλώσω τις προθέσεις μου απερίφραστα. Και ευελπιστώ ότι με το διάλογο που θα έχουμε και όπως είπα και στην αρχή με την εικόνα που σας παρουσίασα για το μέλλον, ελπίζω μετά από την πενταετία θα ε, πιστέψετε και θα το διαπιστώσετε αν με εγκρίνετε ότι, έχω, ότι θα εργαστώ ανεξάρτητα, με διαφάνεια και προς ε, το συμφέρον της Επιτροπής σας αλλά και προς το συμφέρον του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λόρδε Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Σας ευχαριστώ για την ε, θέλησή σας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα να απαντήσετε στις γραπτές ερωτήσεις μας και να επανέλθετε ενώπιόν μας για αυτή τη συμπληρωματική ανταλλαγή απόψεων. Τώρα, αν θέλετε παρακαλώ ε, ένα-δυο λεπτά για μερικές ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ε, ακούσατε και τον κύριο Κατάινεν ε, πριν από μένα. Κάθεστε όλο το πρωί εδώ. Στην τελευταία ερώτηση ε, μου δόθηκε η, ευκαιρία απαντώντας να πω αυτά που ήθελα να πω. Από πλευράς τώρα του χαρακτήρα μου. Ήθελα να σας πω ότι οπωσδήποτε με ενεργητικότητα, ενθουσιασμό και αφοσίωση και ανεξαρτησία βεβαίως θα ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Και βεβαίως ακαιρεότητα. Το μόνο άλλο που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα το τελευταίο εξαήμερο είναι ότι χρειάζεται αντοχή διότι τις τελευταίες εβδομάδες χρειάστηκε πολύ αντοχή χρειάστηκε να υπερβώ κάποιες, ε, κάποια καχυποψία επειδή είμαι Βρετανός και μάλιστα για αυτήν την ε, αρμοδιότητα. Έκανα ό,τι μπορούσα, ελπίζω να καθησύχασα αυτούς τους φόβους παρά τον ε, περίεργο χαρακτήρα του φλερτ μας μέχρι τώρα, ελπίζω να έχω την ευκαιρία από σύντομη σχέση να μετατρέψω τη σχέση μας σε σταθερή και πιο επικερδή. Και ελπίζω να εργαστούμε μαζί για τα θέματα αυτά την προσεχή πενταετία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος για την αντοχή σας, επίσης και για το στυλ σας. Ε, πέρασε τι εδρεγασίε